Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto, ma non credo che sia opportuno fare Καλώς, λοιπόν δεν πρέπει να καθυστερεί ο Αντίπροεδρος και υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Βανάκερε. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με μεγάλη χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας τον σημερινό μας συνομιλητή. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διεύρυνσης είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία μετά τη Λισαβόνα έχει οδηγήσει σε μια αλλαγή θα έλεγα στις εργασίες ε, του Συμβουλίου, γιατί τώρα πλέον έχουμε τον ανώτερο εκπρόσωπο ή είπα το εκπρόσωπο για τα θέματα τα εξωτερικά. Παρ' όλα αυτά η διεύρυνση παραμένει αρμοδιότητα της ε, εναλλασσόμενης Προεδρίας και αυτός είναι ένας λόγος για να συναντηθούμε σήμερα. Πριν λίγες μέρες είχαμε μία συνάντηση με τον Επίτροπο Φούλε Ο Επίτροπος Φούλε ε, μας εξέφεσε τις απόψεις που έχει για τις αρμοδιότητές του. Συγκεντρώσαμε την προσοχή μας λοιπόν σε δύο σενάρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τις συστάσεις και τώρα μένει στο Συμβούλιο να εκφέρει την ε, γνωμοδότηση και να δώσει εντολή στην Επιτροπή πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εξετάζουμε προσεκτικά τις συστάσεις αυτές Υπάρχουν διάφορα σενάρια, διάφοροι υποψήφοι, αυτοί που μπορούν να πλησιάσουν γρήγορα, αυτοί που έχουν εμπόδια. Έχουμε ένα ετερογενές πλαίσιο των χωρών οι οποίες μπορούν να έλθουν κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι πιστεύει το Συμβούλιο λοιπόν γύρω από τα θέματα αυτά. Σας δίνω λοιπόν τον λόγο και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους συναδέλφους. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, χαίρομαι που είμαι μαζί σας σήμερα και που συζητάω μαζί σας μια διαδικασία η οποία ιστορικά βρίσκεται θα έλεγα στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην διαδικασία της διεύρυνσης. Παραδοσιακά οι εναλλασσόμενες προεδρίες το δεύτερο εξάμεινο πρέπει να δώσουν σημασία στο θέμα αυτό περισσότερο από ότι στο πρώτο εξάμεινο γιατί το Δεκέμβριο τα κράτη-μέλη προχωρούν στις αξιολογήσεις των διαδικασιών επί τη βάση των εκθέσεων προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα κάνουμε σε 15 μέρες, τις 14 Δεκεμβρίου δηλαδή εδώ στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό λοιπόν το 2010 δεν είναι εξαίρεση και η Βελγική Προεδρία έχει αναγνωρίσει τις ευθύνες τις οποίες έχει, έχει αναλάβει τις ευθύνες αυτές εν στη διαδικασία και έχουμε χαρακτηρίσει την διεύρυνση σαν μία από τις βασικές προτεραιότητες. Από την 1η Ιουλίου ασχολήθηκα με το θέμα της διεύρυνσης σαν ε, ένας τίμιος διαμεσολαβητής τίμιος διαμεσολαβητής ανάμεσα στους εννέα υποψηφίους και πιθανούς υποψηφίους, αλλά και ε, ανάμεσα φυσικά στα ε, κράτη-μέλη. Όταν πρέπει να είναι κανείς ε, ειλικρινής προς τους υποψηφίους και πιθανούς υποψηφίους, ο τρόπος με τον οποίο θα ενσωματωθούν οι χώρες αυτές εξαρτάται από τις δυνατότητες τις οποίες ανοίγουν και παρέχουν οι διάφορες χώρες και γι' αυτό ο ρόλος μου είναι θα έλεγα να μετριάσω τις προσδοκίες τις οποίες θα πρέπει να έχουν. Και από την άλλη προς τις 27 χώρες μέλη ε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στις 14 Δεκεμβρίου ε, μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση και σαν Προεδρεύων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων βασική μου προτεραιότητα ήταν είναι και θα είναι να σεβαστούμε την εμφάνιση θα έλεγα ενός επίπεδου συνένεσης το οποίο να αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες. Η ετήσια επανάληψη της διαδικασίας αυτής δεν θα πρέπει να μας κάνει να παραγνωρίζουμε την βαθύτατη πολιτική της φύση. Από το 1993 μέχρι το 2007 ο αριθμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξαπλασιαστεί, αλλά με συνθήκες οι οποίες διαφοροποιούνται λόγω της ιστορικής συντηρίας και του επίπεδου βάθους θα έλεγα ολοκλήρωσης που έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες πρέπει να ενσωματώσουν 150.000 κοινοτικής νομοθεσίας, σελίδες εννοώ κοινοτικής νομοθεσίας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι το οποίο επηρεάζει την διαδικασία αυτή, το ότι δηλαδή τώρα έχουμε κλείσει ένα χρόνο από τη συνθήκη της Λισαβόνας, κάτι το οποίο επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει την διαδικασία διεύρυνσης, διατηρώντας πάντα την πορεία προς την ευρωπαϊκή εμβάθυνση και ολοκλήρωση. Νομίζω ότι πρέπει να ορίσουμε σωστά τις συζητήσεις, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι συζητήσεις για τη διεύρυνση ε, στο μέλλον. Βιώνουμε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, καρπό της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης από το 1929, με αυξανόμενα επίπεδα διεθνούς αβεβαιότητας και στις χώρες της Ένωσης και στις υποψήφιες χώρες. Συνεπώς πολλοί αμφισβητούν την χρησιμότητα της διαδικασίας διεύρυνσης. Όπως όμως απέδειξαν τα προηγούμενα κύματα διεύρυνσης, όχι μόνο οι υποψήφιες χώρες ωφελούνται από την είσοδό τους στη μεγαλύτερη ζώνη ελευθέρου εμπορίου, αλλά και η ίδια η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εποφελείται από την ενσωμάτωση των νέων μελών στα πλαίσια της συμπλήρωσης της συμπληρωματικότητας την οποία επιδεικνύει οικονομικά. Πρέπει λοιπόν οι χώρες να συνεισφέρουν και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του 2020 μέσα στο νέο διακανονιστικό πλαίσιο. Πρέπει να ενισχύσουν την εσωτερική αγορά μέσα στην οποία θα ευημερίσουν οι επιχειρήσεις οι κοινοτικές και να ασχοληθούμε επίσης και με τις ανησυχίες που έχουμε σε άλλους τομείς όπως η ασφάλεια, τα διεθνή ε, κλιματικά δίκτυα και τα μεγάλα κενά τα οποία υπάρχουν για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και όταν όλα αυτά γίνουν θα μπορέσουμε να καταστήσουμε την Ήπειρό μας ε, σε όλους τους τομείς ασφαλέστερη από ό,τι στο παρελθόν. Βέβαια όλα αυτά ίσως να μην μπορούν να πείσουν εύκολα την κοινή γνώμη για τα ωφέλη που έχει η διεύρυνση. Η κοινή γνώμη ανησυχεί για την παγκοσμιοποίηση και για προφητείες ευρωπαϊκής παρακμής. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι κλειδί για να υπάρξει μια συνένεση στον τομέα της διεύρυνσης όπως υπόθηκε για πρώτη φορά το 2006. Καταρχάς, η κοινή γνώμη αλλάζει πολλές φορές άποψη και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες και να εξηγήσουν σωστά τις ευκαιρίες που ανοίγει η διεύρυνση. Και δεύτερον, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας της διεύρυνσης. Από πλευράς κρατών μελών σημαίνει ότι πρέπει να αμείβουμε την πρόοδο μια χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την παρέμβαση διμερών θεμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα κάθε υποψήφια χώρα μπορεί να μπει στην Ένωση μόνο όταν αντικειμενικά είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη του μέλους. Αυτό σημαίνει για τις υποψήφιες χώρες. Πρώτον, από το να μην δίνουν ε, θα έλεγα υποσχέσεις προς τους πληθυσμούς τους που δεν μπορούν να κρατήσουν και δεύτερον να δημιουργούν ένα κλίμα οι υποψήφιες χώρες το οποίο να είναι θετικό σε περιφερειακές συγκρούσεις. Όλες αυτές οι αρχές έχουν επιβεβαιωθεί και ε, θα έλεγα διευκρινιστεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2006. Νομίζω ότι ο σεβασμός αυτών των βασικών αρχών είναι η μοναδική εγγύηση για την μακροπρόθεσμη διάρκεια θα έλεγα και ταυτόχρονα αξιοπιστία του συστήματος της διεύρυνσης τα, ε, οι εμπειρίες που έχουμε συλλέξει στον τομέα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι κάτι το θετικό. Εφόσον βάζουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ταυτόχρονα δώσουμε τα ωφέλη όπως οι βίζες, αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα και για μας και για τις υποψήφιες χώρες. Επιτρέψτε μου τώρα κυρίες και κύριοι να επανέλθω λίγο στην πρόοδο που συντελέστηκε τους τελευταίους 12 μήνες από τις εννέα υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες που έκαναν τη στρατηγική επιλογή της κοινοτικής προοπτικής. Να ξεκινήσω με την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μαυροβούνιο και την Αλβανία και για τις δύο χώρες. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις θετικές εξελίξεις. Συστήνει όμως οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν μετά από την επίτευξη περαιτέρω σημαντικών προτεραιοτήτων. Για το Μαυροβούνιο, στα πλαίσια της προόδου της ουσιαστικής που έχει επιτελεστεί, διαπιστώνουμε κενά, αλλά παρόλα αυτά συστήνουμε να χαρακτηριστεί η χώρα αυτή υποψηφία τον Δεκέμβριο. Παρόλα αυτά, για να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις πρέπει να πετύχουν 7 επίπεδα νέων προϋποθέσεων, ε, κράτος δικαίου, ελευθερία μέσων ενημέρωσης, εκλογική μεταρρύθμιση, καταπολέμηση διαφθοράς και καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος. Για την Αλβανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη πολλαπλασιασμού των προσπαθειών πριν δοθεί στη χώρα ο χαρακτηρισμός υποψηφία χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, όταν υπάρξει μια περαιτέρω θετική αξιολόγηση της προόδου της συγκεκριμένης χώρας. Θα πρέπει να προωθηθεί ο διάλογος ανάμεσα στα αλβανικά πολιτικά κόμματα μετά από τις εκλογές του 2009. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο και δεν ε, ε, εκπλήσεται κανείς ότι όπως είχα πει και τον Οκτώβριο, ε, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι επαφές αυτές είναι η εύρυθμη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος στην χώρα αυτή. Βέβαια έχει υπάρξει πρόοδος ε, και έχει αναφερθεί στα βήματα που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κράτος δικαίου, καταπολέμηση διαφθοράς κτλ να στραφώ τώρα στις υποψήφιες χώρες που έχουν το όνομα της υποψηφίας δηλαδή. Ε, Κροατία ξεκινώ, οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν στην τελική φάση με 33 από τα 35 κεφάλαια του κεκτημένου ανοιχτά και 22 από αυτά προσωρινά κλειστά. Εφόσον τα λεγόμενα benchmarks ε, ε, θα έλεγα κατακτηθούν, τότε οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στις 22 Δεκεμβρίου τη ευκαιρία της ε, τρίτης ενταξιακής διάσκεψης με την Κροατία. Και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η διατύπωση της συνθήκης προσχώρησης όπως ζητήθηκε από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2009. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς. Παρ' όλα αυτά η Κροατία απαιτείται να προχωρήσει σε πληρέστερη συνεργασία με το Διεθνές Δικαστήριο για την Τέος Γιουκοσλαβία, εντατικοποιώντας τις προσπάθειες που κάνει για να ικανοποιήσει τις απαιτήσει της, της ε, Διεθνούς Εισαγγελίας για έγγραφα στρατιωτικής φύσεως. Πολλά μένει να γίνουν και στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού, όπως επίσης και στον τομέα του δικαστικού σώματος και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η έκθεση παρακολούθησης της εξέλιξης της κατάστασης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δικαστικής εξουσίας των στις 11 Μαρτίου του 2011 θα είναι ένα περαιτέρω μέτρο για να πιεστεί θα έλεγα η Κροατία έτσι ώστε την ημερομηνία ένταξης να έχει κάνει όλα τα απαιτούμενα βήματα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της Τουρκίας. Η Τουρκία συνέχισε τη διαδικασία πολιτικής μεταρρύθμισης. Παραμένουν ανησυχίες για την ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης, γενικότερα έκφρασης, όπως επίσης και για τα γενικότερα δικαιώματα και τα μειονοτικά δικαιώματα, και ε, υπάρχει μόνο επιμέρους εφαρμογή του δημοκρατικού ανοίγματο σχετικά με το κουρδικό. Επαναλαμβάνοντας βέβαια την πλήρη καταδίκη των τρομοκρατικών ενεργειών την οποία είπα στην Άγκυρα ε, το καλοκαίρι, επαναλαμβάνω την έκφραση αλληλεγγύης προς τα θύματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι περιμένουμε και από πλευράς της τουρκικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το κουρδικό συνολικά. Πέραν αυτού, αν και πρέπει πολλά να γίνουν ακόμα, το πακέτο συνταγματικών τροπολογιών, το οποίο ενεκρίθη από το δημοψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου, είναι ένα θετικό βήμα. Η ξεκάθαρη λαϊκή υποστήριξη που έδωσαν οι Τούρκοι πολίτες για την περαιτέρω ενίσχυση των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου στη χώρα τους είναι κάτι το οποίο απαιτεί δύο περαιτέρω ενέργειες, δύο περαιτέρω στοιχεία. Πρώτον, την εφαρμογή του πακέτου σύμφωνα με τα κοινωνικά στάνταρτς, σχετικά δηλαδή με τις εφαρμοστικές διατάξεις των αλλαγών της μεταρρύθμισης και δεύτερον, μια συνολικότερη συμμετοχή ε, που θα οδηγήσει ε, τους ενδιαφερομένους σε νέες προτάσεις για περαιτέρω συνταγματικές αλλαγές. Υποτίθεται ότι εδώ έχουμε την υποχρέωση του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος την επόμενη άνοιξη θα κάνει προτάσεις για διορθώσεις στο Σύνταγμα το οποίο είχε γίνει δεκτό κάποτε επί στρατιωτικής δικτατορίας. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στη χώρα αυτή το καλοκαίρι και με τη συμμετοχή μου στη διάσκεψη του Βοσπόρου τον Οκτώβριο, απίθυνα έκκληση στους Τούρκους συνομιλητές μου για την πλήρη εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλου στη Συμφωνία Σύνδεσης. Σχετικά με την επανένωση της Κύπρου. Δεν ήθελα εγώ να ανοίξω μια παράλληλη διαδικασία για το κυπριακό ευρωπαϊκού τύπου, αλλά σεβόμενοι τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευκολύνουμε την, τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ξέρετε ότι το πράσινη βίβλο για την ενημέρωση από πλευράς εμπειρογνωμόνων και την επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων στην Άγκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις από την Τουρκία σε σχέση με τα κεφάλαια τα οποία δεν έχουν κλείσει και ίσως το Συμβούλιο να μην είναι σε θέση να ξεκινήσει νέα κεφάλαια αυτό το εξάμεινο. Αν κάτι τέτοιο σημαίνει ε, ότι θα, αν κάτι τέτοιο συμβεί μάλλον, αυτό θα σημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ξυπνητήρι, σαν προειδοποίηση για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Με ξεκάθαρο τρόπο θα ήθελα να πω ότι η Βελγική Προεδρία συνεχίζει μέχρι και την τελευταία μέρα της προσπάθειές της έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρία θα έλεγα για να σημειωθεί η πρόοδος στο Κυπριακό. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2005 της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκκίνηση διαπραγματεύσεων που θα είναι επωφελής και για την Τουρκία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ισλανδία Προείδρευσα της ε, πρώτης διάσκεψης σχετικά με το θέμα της, πρόσβα... της ε, ε, Ισλανδίας και όπως είπα και στον συνάδελφό μου από την χώρα της Ισλανδίας, οι στενές σχέσεις της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας για την ικατοποίηση των κοινοτικών στάνταρ θα βοηθήσει τη διαδικασίε ένταξης. Παρ' όλα αυτά η Ισλανδία θα πρέπει να ενσωματώσει πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο και στον τομέα της αλληλείας και στον τομέα της φαλενοφυρίας και να σεβαστεί όλες τις συμφωνίες της ευρύτερης ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης όπως τον τομέα σαν παράδειγμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Δεν θα έχουμε αποτελέσματα από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από τα θέματα αυτά πριν από τα μέσα του 2011. Σχετικά με τη ΦΥΡΟΜ, έχει υπάρξει πρόοδος, αν και με άνισο ρυθμό σε σχέση με το παρελθόν, στον τομέα των μεταρρυθμίσεων του Κοινοβουλίου, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, του δικαστικού σώματος, της δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου. Ξέρετε ότι είχε ληφθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2009, αλλά ξέρετε ότι απαιτείται μια ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για να ξεκινήσουν πραγματικά οι διαπραγματεύσεις. Όπως είπα στον συνάδελφό μου Αντώνιο Μιλοσόσκη όταν προείδρευσα του Συμβουλίου Σύνδεσης τον Ιούλιο, μία θέση, μία λύση μάλλον του προβλήματος ε, του ονόματος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών είναι κάτι το θεμελιώδες. Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση στα Σκόπια θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας. Θα κλείσω κύριε Πρόεδρε με τρεις υποψήφιες δυνητικά ε, χώρες. Λοιπόν, Σερβία, ξέρετε ότι η Προεδρία η Βελγική ε, διευκόλυνε την επίτευξη συνένεσης στο Συμβούλιο έτσι ώστε να υποβάλει η, έκθεση, η Επιτροπή την έκθεσή της για τη Σερβία λέμε ότι η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι προϋπόθεση για να γίνει μέλος και φυσικά είναι κρίσιμο το θέμα της σύλληψης των δύο τελευταίων ε, καταζητουμένων. Σχετικά τώρα με την μεταρρύθμιση του δικαστικού πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την εκρίζωση των προβλημάτων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Σε περιφερειακό επίπεδο συνεχάριν τον πρόεδρο Τάντιτς για τα σημαντικά βήματα που έκανε για τη συμφιλίωση των ναών και των χωρών της περιοχής προς την Βοσνία Ερζεγοβίνη και σχετικά με το τραγικό θα έλεγα αποτέλεσμα της κληρονομιάς της Ρεμπρένιτσα Υπάρχει ένα ψήφισμα λοιπόν που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τη Σερβία με την αιγίδα θα έλεγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που πιέζει προς τον διάλογο Βελιγραδίου-Πριστίνα. Ο διάλογος αυτός θέλουμε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν. Μετά για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετά από την σωστή διεξαγωγή των εκλογών του Οκτωβρίου και 15 χρόνια μετά από τις συμφωνίες της ειρηνευτικές του Ντέιτον, οι πολίτες της Βοσνίας Ευζεγοβίνης ε, αξίζουν ένα ποιοτικό βήμα ε, προς τα εμπρός, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν συναντήθηκα με τον συνάδελφο Αλ Καλάη τον προηγούμενο μήνα, αυτό είναι το μήνυμα που του ζήτησα να μεταφέρει σε όλους τους πολιτικούς του εταίρους στην πορεία για την ευρωπαϊκή προοπτική οι κοινότητες της χώρας θα πρέπει να βρούνε τις κοινέ μεθόδους για την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Προσαρμογή του συντάγματος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και ε, φυσικά εφαρμογή σωστή του κοινοτικού κεκτημένου και ε, επίσης προϋποθέσεις σχετικά με το κλείσιμο του γραφείου του υπάτου εκπροσώπου. Τώρα, για το κοσιφοπέδιο. Θετικά στοιχεία ήταν η αποκέντρωση, όπως επίσης και οι ε, δημοτικές εκλογές στις σερβικές περιοχές του κοσιφοπεδίου και καλύτερη συμμετοχή με την αποστολή Γιούλεξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά παραμένουν σοβαρές ανησυχίες στον τομέα του κράτους δικαίου, σε σχέση με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της έκπληξης βρώμικου χρήματος. Υπάρχει εδώ το θέμα και της αναγνώρισης της συγκεκριμένης χώρας σε σχέση με το καθεστώς της συγκεκριμένης χώρας. Ε, η Επιτροπή ζητά να υποστηριχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως του Κωσυφοπεδίου και αυτό είναι κάτι το θετικό. Τα μέτρα αυτά βρίσκονται υποσυζήτηση από τα κράτη-μέλη και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια υπογραφή μελλοντική εμπορικής συμφωνίας και ένα διάλογο για τη χορήγηση θεωρήσεων στα πλαίσια επίσης και της προόδου στον τομέα των, των προσφύγων που επιστρέφουν στη χώρα. Στα πλαίσια του διαλόγου <coughs> με το Βελιγράδι δεν θα ξεχαστεί η ευρωπαϊκή προεπτική. Τελειώνοντας με τα Δυτικά Βαλκάνια, Αναφέρομαι στις κοινέ προοπτικές χωρών οι οποίες ήταν εμπόλεμες πριν λίγα χρόνια. Και αυτό δείχνει ε, τι χρήσιμο αντιπροσωπεύει το ευρωπαϊκό θα έλεγα ιδεώδες εδώ και αρκετά χρόνια. Η επιθυμία των λαών για την ειρήνη και τη σταθερότητα είναι δεδομένη. Αυτή η ειρήνη θα έλεγα οδηγεί σε μια κοινή ευημερία χωρίς να λυθούν βέβαια όλα τα επιμέρους περιφερειακά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά έχει υπάρξει πολύ σημαντικά βελτιωμένη περιφερειακή συνεργασία, κάτι το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τις εντάσεις που σοβούν στην περιοχή. Κάποιες ε, εξελίξεις έχουν υπάρξει στον τομέα της διεύρυνσης, ε, οι οποίες ε, μπορεί, εφόσον δεν δείξουν τα εμπλεκόμενα μέρη την απαιτούμενη πολιτική βούληση για να ξεφύγουν από το αδιέξοδο, να επιβαρύνουν την κατάσταση αλλά εφόσον διατηρηθεί η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εφόσον εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει τη διαδικασία, τότε θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ε, στην μελλοντική ευημερία των χωρών αυτών, ενισχύοντας τις περιφερειακές μορφές συνεργασίας. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ξεκινάει η συζήτηση. Σαλαφράγκα. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Προεδρεύοντα. Σας ευχαριστώ για την γενική επισκόπηση που μας κάνατε για τις υποψήφιες για ένταξη χώρες ή τις δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες υπό το φως της έκθεσης πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά περιμένουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών. Συμφωνώ μαζί σας ότι κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να κρίνεται αξιοκρατικά, αλλά και υπό το φως των ιδιαίτερων συνθήκων. Και η πολιτική βούληση είναι με απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά όχι και επαρκής. Και ακόμη και αν είναι συγκυριακές οι προσωρινές ε, συνθήκες, ε, θα πρέπει και αυτές να τις λαμβάνουμε υπόψη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, Πρώτον, μια ναι, και πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο όραμα και μακροπρόθεσμη προοπτική. Συνεργάζεστε με την προηγούμενη και την επόμενη Προεδρία. Έχετε στενή συνεργασία ε, οι τρεις διαδοχικές Προεδρίες. Ως προς τις ε, περιστάσεις, μας είπατε ότι την 1η Δεκεμβρίου εορτάσαμε την πρώτη επέτειο τη θέσεις εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, που έδωσε και την όθηση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που επειδή καθυστέρησαν οι διαπραγματεύσεις, ε, τέθηκε σε εφαρμογή κάπως αργότερα. Δεν εξελέγει βέβαια ο Λουί Μισελ, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ε, δυτικό μπλοκ υποστήριξε ε, άλλον υποψήφιο. Επίσης ε, είχαμε το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου στην ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ερωτώ λοιπόν, η όθηση που κανονικά θα έπρεπε να είχε δώσει η συνθήκη της Λισαβόνας χαρακτηρίζει και την διαδικασία διεύρυνσης ή μήπω επικρατεί μια δράνεια και δεν υπάρχει καμία ποιοτική αλλαγή. Μας κάνετε μια λεπτομεριακή ανάλυση για την κάθε υποψήφια χώρα υπό το φως της σοβούσας οικονομικής κρίσης. Τι κλίμα επικρατεί στο Συμβούλιο για τη διεύρυνση. Είπατε ότι δίνετε προτεραιότητα σε αυτή την ενταξιακή διαδικασία. Εστερνίζετε το Συμβούλιο αυτή την προτεραιότητα ή εξαιτία τη ε, της οικονομικής και της χρηματοπιστωτικής κρίσης θα, θα συνεχίσουμε ε, σαν να μην συνέβαινε τίποτα ιδιαίτερο και ή αντίθετα θα δοθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μια νέα όθηση στην ενταξιακή διαδικασία και στη διεύρυνση. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Φλότρ, που είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον ε, Βέλγο Υπουργό για την παρουσίαση. Συμφωνώ μαζί σας ότι η διαδικασία της διεύρυνσης είναι μια ιδιαίτερα πολιτική διαδικασία και πολλές φορές είναι και εξαιρετικά ευαίσθητη. Ως προς την Τουρκία θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε τα περισσότερα επιχειρήματα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, για παράδειγμα, για να επιβραδύνουν ή να θέσουν υποδιαφορετική προοπτική τις ενταξιακές διαδικασίες το ποσοστό ανάπτυξης Τουρκίας ε, και η εύρωστη αγορά απασχόλησης ε, ε, θα μπορούσε να, να την, θα μπορούσε να την υποφθαλμίουν πολύ εδώ στην Ευρώπη. Αλλά εγώ προτιμώ μια βιώσιμη περισσότερη ανάπτυξη, μια υφόρο οικονομική ανάπτυξη. Αυτά τα λέω για να αποδείξω ότι η οικονομική και η πολιτική κατάσταση δεν είναι πάντα αρνητική προϋπόθεση ή μάλλον δεν δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία της διεύρυνσης. Είπατε ότι θα εθαρρύνεται τη διαδικασία στην Τουρκία για την συνταγματική αναθεώρηση, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Και αυτό διαπιστώνουμε και οι ευρωβουλευτές όταν πηγαίνουμε στην Τουρκία. Θέλουμε την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Να είμαστε αποφασιστικοί και μονοσήμαντη σε αυτά τα μηνύματά μας. Εσείς πάντως, τι μήνυμα σκοπεύετε να μεταφέρετε στο Συμβούλιο, στα μέλη του Συμβουλίου, ως προς την Τουρκία. Γιατί εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ενία μηνύματα προς την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε τη στρατηγική μας, τους στόχους μας και την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας που εφαρμόζουμε στο Συμβούλιο. Γιατί θα ήταν απογοητευτικό, για να μην πω ανησυχητικό, στη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας, στη διάρκεια της Προεδρίας δηλαδή μιας χώρας που έδειξε μεγάλη πολιτική βούληση να υποστηρίξει την διαδικασία της διεύρυνσης. Για πρώτη φορά στη διάρκεια μιας προεδρίας να μην ανοίξει κανένα κεφάλαιο διαπραγμάτευσης για ένα ολόκληρο εξάμεινο. Παρά τις νομοθετικές ε, μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Τουρκία και που επιτρέπουν ε, το άνοιγμα του κεφαλαίου για τον ανταγωνισμό, για παράδειγμα. Ερωτώ λοιπόν, εσείς στο Συμβούλιο τι μηνύματα θα δώσετε στις προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να δώσουμε το μήνυμα για μια αξιόπιστη, σαφή, συνεπή διαδικασία που θα είναι δίκαιη και θα σέβεται και τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Γιατί οι αφιβολίες ε, που επικρατούν μερικές φορές είναι ολέθριες για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, αλλά και για την επιτυχία της, ε, διαδικασίας εκδημοκρατισμού της Τουρκίας. Καλό θα ήταν ε, η Βελική Προεδρία να αναλάβει κάποιες προεδρίες για να ξεφύγουμε αυτή την κόπωση που φέρνει σε αποτελμάτωση την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας. Ο κύριος Κάτσιν, που είναι ο εισηγητής μας για τη Σερβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προσπάθειες κάνετε εσείς για να προχωρήσει η κατάσταση εντός της Κύπρου. Δεν μιλάω για την Τουρκία και τη στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις των δύο προέδρων για να ξεπεραστεί η παρούσα κατάσταση και για να γίνει δυνατή κάποια στιγμή στο μέλλον η επανένωση του νησιού. Εσείς, ε, η Βελική Προεδρία, είστε έτοιμοι να αναλάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία πριν το πέρας το εξαμήνου σας. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα βασικά να κάνω τρεις ερωτήσεις ε, ε στο Προεδρείο, στον ε, Υπουργό Εξωτερικών της, ε, του Βελγίου. Ο κύριος υπουργό μας ε, μίλησε για ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά τη Συμφωνία της Οχρίδας στην πρώην Οικοσταβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μάλιστα είπε η ανάγκη να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία. Μπορεί να μας εξηγήσει σε τι συγκεκριμένα αναφέρεται, ποιες είναι οι ανησυχίες του κύριου Υπουργού. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ένα δεύτερο ζήτημα που ήθελα να τον ρωτήσω, δεν έγινε κατανοητή ερώτηση νομίζω. Ε, ένα δεύτερο ερώτημα entendu Σας άκουσα, αλλά μιλάτε για μια συμφωνία. Συμφωνία, εγώ δεν είπα συμφωνία. Si Είχα καταλάβει ότι αναφερόσα στην ε, συμφωνία της Οχρίδας. Και ποια είναι η ερώτηση σας ακριβώς? Έχετε κάποια ανησυχία αυτής της ε, συνθήκης. Υπάρχουν ζητήματα που σας ανησυχούν, δεν εφαρμόζονται. Ποια είναι αυτά. Ε, η δεύτερη ερώτηση αφορά την Κροατία. Διάβασα ε, ότι σε μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία των Κροατών που είναι αντίθετη στην ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους ισχύει αυτό το πράγμα και ποιες είναι οι συνέπειες, αν, αν σας είναι γνωστές. Και ένα τελευταίο ζήτημα ε, αφορά ε, τις εξελίξεις στη Βοσνία-Ζεγοβίνη και το θέμα του, του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας αν υπάρχουν του ΟΗΕΝΟ, αν υπάρχουν κάποιες προοπτικές και πότε για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Και η τελευταία τελευταία ερώτησή μου αφορά το καθεστώς του Κωσόβου. Υπάρχουν ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Συμβουλίου, σε επίπεδο των ευρωπαϊκών ε, οργάνων, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης του Κωσόβου από τις χώρες οι οποίες ακόμα δεν το έχουν αναγνωρίσει. Αυτά. Σας ευχαριστούμε κύριε Αγκουράκη. Το λόγο έχει ο κύριος Πόσελτ. Äh, um Πρόεδρε, έχουμε έρθει εδώ για να μάθουμε καινούργια πράγματα. Γι' αυτό έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα ολοκληρωθούν κάποια από τα κεφάλαια με την Κροατία και αν ναι, πόσα. Και πιστεύετε ότι υπό Ουγγρική Προεδρία θα μπορούν να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Σκοπεύετε το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο να επιβάλλετε η Μακεδονία να λάβει μία ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων το επόμενο έτος. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες μου ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πόσα. Ο κύριος, η κυρία κορνέλη έχει το λόγο. Yeah, you. Um, a few... Ευχαριστώ. Έχω παρατηρήσεις ε, για τη Βοσνία, τη Μακεδονία και το Διεθνές Δικαστήριο, Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία. Για τη Βοσνία είπατε ότι θα πρέπει οι πολιτικοί να βρουν ένα κοινό έδαφο συνεννόηση. Δίκιο έχετε. Αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να βρουν ένα κοινό έδαφο και να εθετήσουν ε, μια θέση στεναρή. Υπάρχει, υπάρχουν πολλές διαφωνίες αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν ε, προτάσεις για κλείσιμο του γραφείου της ΥΠΑ της και ε, στη Βοσνία πολλοί λένε ότι οι διεθνείς αποστολές θέλουν να εγκαταλείψουν τη Βοσνία το συντομότερο δυνατόν. Ενώ το αντίθετο μήνυμα θα πρέπει να στείλουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τη Βοσνία και δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουμε αν δεν υπάρχει ένα ενωμένο ομοσπονδιακό κράτος. Και θα χρειαστεί διεθνής παρουσία εκεί μέχρι να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα πρέπει να καλέσουμε την Λέδη ε, Άστον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν ε, πρωτοβουλία για μια καλά προετοιμασμένη μεταρρυθμιστική διαδικασία που θα οδηγήσει και σε νέο σύνταγμα στη Βοσνία. Υπάρχουν καθόλου εξέλιξει σχετικά για τη Σερβία. Η απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου αναφέρει ότι το Συμβούλιο θα προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια είναι απαραίτητη στη Σερβία για τη σύλληψη των φυγοδίκων Χάτζης και Μλάντιτς. Πολύ καλή ιδέα και θα πρέπει όντως να δραστηριοποιηθεί το Συμβούλιο και να ε, βοηθήσει τη Σερβία με, με τεχνογνωσία ή με οικονομικά μέσα για να συλλάβει το συντομότερο τους φυγάδες. Και τέλος για τη Μακεδονία. Την τελευταία φορά που συνομίλησα με εκπροσώπους της Μακεδονίας, διαπίστωσα ότι φθήνει όλο και περισσότερο στα μάτια τους η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα αυτή αισθάνεται ότι υπόκειται εκβιασμό από μια χώρα που είναι ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι σε μια χώρα που ε, δεν είναι και υπάρχει ένας πολύ άνισος συσχετισμός δυνάμεων το Συμβούλιο θα επιληφθεί αυτής της κατάστασης ή θα ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα για να αποσυνδεθεί το ζήτημα της ονομασίας από την πρόοδο της Μακεδονίας για ένταξη. Γιατί με βάση την πρόοδο που έκανε η χώρα αυτή αξίζει η προώθηση της ενταξιακής της προοπτικής. Σας ευχαριστούμε κυρία Κορνέλισεν. Ο κύριος Σέψλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, ε, τι, ε, ε, ποιο θα είναι το κληροδότημα που θα αφήσετε στην Ουγγρική Προεδρία, πώς, ε, πόσο αποτελεσματική πιστεύετε ότι θα είναι, έχετε κάποιες συστάσεις προς την επερχόμενη Προεδρία και τι εμπειρίες είχατε από τη, από τη συνεργασία των τριών ε, διαδοχικών προεδριών. Αναφερθήκατε στο καθήκον που έχουν κυβερνήσεις προς το λαό τους. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και πολλοί προσπαθούν να το αποφύγουν. Πάντως ο Ευρωπαϊκός Δήμος, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος, καλό θα ήταν να μπορεί να έχει λόγο για τη διεύρυνση. Όταν μιλούμε για διεύρυνση, δεν είναι ότι μπαίνει απλώ μια νέα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι διευρύνεται ο Ευρωπαϊκό Δήμο. Αυτό το θέμα πώ θα το αντιμετωπίσετε, πώ θα το λύσετε. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο. Α, συγγνώμη, κυρία Λούνατσεκ. και μετά ο κύριο Στάνοκ. Η κυρία Λούνατσεκ και μετά ο κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω. Στίβεν, ακόμη καλύτερα. Πολύ ευχαρίστως και πολύ ευκολότερα. Γεια σου, Στίβεν. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχα συνάντηση με εκπροσώπους Αρμενίας, ε, οπότε έπρεπε να φύγω και από εκεί. Ε, πήγα πέντε μέρες στο Κωσυφοπαίδιο, λίγο πριν τις εκλογές και είμαι εισηγήτρια για το Κωσυφοπαίδιο. Έχω μία ερώτηση για το Κωσυφοπαίδιο λοιπόν. Την ε, έθεσε και ο προλαλής σας και εγώ όπως και ο συνάδελφος θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει καμία πρόοδος ότι αφορά την αναγνώριση του Κωσυφοπαιδίου από τις πέντε χώρες που δεν το έκαναν ακόμη, δεν, την, δεν προέβησαν στην αναγνώριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διάφορα θεσμικά της όργανα και τις αποστολές που έχει επιτόπου δεν έχει να επιδείξει μια ενιαία συσπηρωμένη θέση, ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει μια ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διαρωτώνται ότι η αποτελμάτωση ε, στο διάλογο για τις θεωρήσεις ε, σχετίζεται με το γεγονός ότι πέντε χώρες δεν αναγνώρισαν, ε, γιατί δίνεται προνόμιο στη Σερβία και προωθείται περισσότερο η δική της πορεία εις βάρος του κοσυφοπεδίου. Υπάρχει καμία πρόοδο στο θέμα της αναγνώρισης του κοσυφοπεδίου και επίσης το θέμα των, της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για το κοσυφοπέδιο. Οι Αλβανοί, οι Βόσνοι έχουν από τις 15 Σεπτεμβρίου, από τις 15 Δεκεμβρίου αυτή τη δυνατότητα. Η, ο μοναδικός λαός που περιθωριοποιήθηκε, που αισθάνεται απομονωμένος ε, και οι νέοι ε, που έχουν μείνει στο περιθώριο είναι οι νέοι του Δεν μπορούν να, να κυκλοφορήσουν χωρίς ε, θεωρήσει και να δουν τι θα πει η Ευρώπη. Επίσης, ε, καλό θα ήταν να ενισχύσουμε τις πολιτικές δυνάμεις του κοσυφοπεδίου. Υπάρχει ένα κόμμα που θέλει αυτοδιάθεση και θέλει να διώξει όλους τους ξένους παράγοντες στο κοσυφοπέδιο και επίσης από ό,τι ξέρω και στο Συμβούλιο υπάρχει απροθυμία ως προς την πρόθεση του διαλόγου για τις θεωρήσεις τουλάχιστον. Να ξεκινήσει ο διάλογος για τις θεωρήσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστια απογοήτευση και εκνευρισμό στο λαό του Κωσυφοπεδίου και εξαιτία αυτού του θέματος χάνουμε την υποστήριξη του λαού για την ενταξιακή προοπτική της χώρας αυτής. Πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη ότι το Κόσοβο και οι Κωσοβάροι θα πρέπει ήδη από τώρα να εμπλακούν στον διάλογο για τις θεωρήσεις. Τώρα, όχι από αύριο. Δεύτερο ερώτημα για το Μαυροβούνιο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ιδιωτικοποίηση σε θέματα ενεργειακά, γιατί η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου είναι γνωστή για την αδιαφάνειά της, για να το πω κατεφημισμών. Πώς θα αυξηθεί η διαφάνεια λοιπόν σε, στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Κάνετε κάποια προσπάθεια για περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη διαφθορά και δωροδοκία στο Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εγώ είμαι ο εισηγητής για το Μαυροβούνιο, αλλά δεν θα μιλήσω για το Μαυροβούνιο, γιατί δεν είναι επίμαχο το θέμα του Μαυροβουνίου. Γι' αυτό και είναι ανακούφιση για μένα που έχω το Μαυροβούνιο και όχι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Πάντω, ε, μετά από αυτά που είπε η κυρία Λούνατζεκ, φαντάζομαι και η ομάδα τη και η ίδια θα υποβάλει τροπολογίε. Πάντω, για την ιδιωτικοποίηση, συμφωνώ ότι καλό θα είναι να γίνει με σωστό και διαφανή τρόπο. Και χαίρομαι που θα ιδιωτικοποιήσουν ε, τομείς που παραδοσιακά ελέγχονταν από το κράτος. Έχω μία πιο γενική ερώτηση σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πώς λειτουργήσε στην πράξη η εκπεριτροπής Προεδρία και τι εμπειρία είχατε εσείς ως Υπουργός Εξωτερικών μετά την ενίσχυση της εξωτερικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την παρουσία δηλαδή της κυρίας Άστον, αντιπρόεδρο της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου, του κ. Βαν Ρομπόη. Ποιο είναι ο ρόλο τη κάθε σα, Υπάρχει καλή, καλός συνδυασμός και συνάρθρωση και η, η, πώς η εναλλακτική προεδρία αυτή, η διαδοχική προεδρία θα είναι πλέον κάτι, ένα ιστορικό απομεινάρι και θα είστε η τελευταία προεδρία που θα έχετε πως ουσιαστικό έργο και όλες αυτές οι προεδρίες θα εξαφανιστούν οι εκπεριτροπής όταν θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όταν η ΚΕΠΑ γίνει κάτι πιο σταθερό. Θα χαθεί πιο ρόλο της εξάμεινε εκπεριτροπής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κασουλίδης είναι ο τελευταίος ομιλητής. Chairman, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι είσαστε ένας τίμιος διαμεσολαβητής προσπαθώντας να βρείτε λύσεις στα θέματα του πρωτοκόλλου της άκρας και κάποια από τα κεφάλαια που ε, είναι αντικείμενα διαπραγματεύσεων. Μπορείτε να ενημερώσετε την Επιτροπή μας ε, όσον αφορά τις συγκεκριμένες σας προσπάθειες. Αν όχι, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι εδώ αυτό που είπατε, δηλαδή η απόλυτη εφαρμογή χωρίς διακρίσεις του πρωτοκόλλου της Άγκυρας είναι αυτό που σκοπεύετε να κάνετε. Σε ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. Εσείς κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο. Έχετε δέκα παρεμβάσεις και πολύ περισσότερο ρωτήσεις να απαντήσετε. Ναι. Θα προσπαθείτε είμαι πλήρης στις απαντήσεις μου, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα σχόλια που έγιναν και σημείωσα και τα περισσότερα σχόλια που έχουν σε στόχο μάλλον ε, να ακουστούν κάποια μηνύματα ίσως και δεν ήταν ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω Να απαντήσω πάντως. Ο κύριος Σαλαφράγκα που αναφέρθηκε σε κάποιες από τις πρόσφατες εξελίξεις για το ότι έγινε σε κάποιες πληροφορίες στα Ηνωμένα Έθνη βρίσκεται πιο μακριά από αυτή καθ' αυτή την διαδικασία διεύρυνσης. Είναι αληθές ότι αν η συνθήκη της Λισαβόνας μας θέτει στην δυνατότητα να μιλήσουμε με μία φωνή, αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο για λόγια αλλά και για την πράξη. Έχετε δίκιο. Ο κύριος Αλαφράγκα αναφέρθηκε στη λεγόμενη κόπωση διεύνησης. και απαντώντας αυτά και σε κάποιες από τις ε, άλλες απαντήσεις θα ήθελα να πω ότι Εμεί εξετάσαμε προσεκτικά το θέμα του ορίζοντα 31 του 2010 γιατί ξέραμε ότι δηλώσεις είναι άχρηστες εάν δεν ακολουθούν από συγκεκριμένες πράξεις. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε με το σκεπτικό ότι θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται το τρένο. Κάποιοι είπαν ότι θα πρέπει να είναι μια δίκαια διαδικασία. Δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά όλες οι χώρες, να το έχουν υπόψη, τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, αλλά να αντιδράμε ανάλογα με τις ανάγκες. Ξανατονίζω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία δεν βασίζεται ε, σε ένα χρονοδιαγράμμα. Είναι σαν ένα φοιτητή που λέει πότε θα έχω το δίπλωμά μου σαν φοιτητή μπορεί να ρωτήσει κανένα πότε θα έχω εξετάσει. Αλλά πότε θα έχω το δίπλωμα εξαρτάται το πώ έχει δουλέψει. Και εδώ το ίδιο έχουμε πρέπει να δουλέψουν και να ενσωματώσουν το κοινοτικό και εκτιμένο. Να πούμε λοιπόν ότι συνεχίζουν να κινούνται. Δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε την κατάσταση αλλά αυτή δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να βασιστεί σε ένα σκεπτικό χρονοδιαγράμματος. Όταν είπε η κυρία Φλότρο ότι δεν είναι αρνητικό το περιβάλλον λόγω των οικονομικών αναγκαιοτήτων, έχει δίκιο και θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα επίσης ότι η διαδικασία διεύρυνσης η οποία από πολλούς θεωρείται σαν απειλητική προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να έχει κανένας την τόλμη να το πει. Και όταν με ρωτάτε λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα που μεταβιβάζω στους συναδέλφους στο Συμβούλιο, ακριβώς αυτό. Ιδίως το παράδειγμα που αναφέρατε, στη χώρα στην οποία αναφερθήκατε, στην Τουρκία δηλαδή, αυτό που πρέπει να κοινοποιήσουμε στους 26 συναδέλφους ε, στο Συμβούλιο είναι ότι σε μια σειρά επισκέψεων τους τελευταίους μήνες στην Τουρκία μίλησα με πολλούς εκπροσώπους παραδείγματος χάνει θρησκευτικών μειονοτήτων, πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικονομικούς ε, κύκλους που δεν σχετίζονται άμεσα με το κυβερνόν κόμμα, μάλλον πιο επικριτική είναι προς το κυβερνόν κόμμα. Και κάθε μία από τις πηγές που χρησιμοποίησα τονίζει ότι πολλές από τις τροποποιήσεις και οι αλλαγές που έγιναν στην Τουρκία οφείλονται ακριβώς σε αυτή την ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Και μου είπανε, σας παρακαλούμε, φροντίστε να μην στρέψει τα νότα της προς την Τουρκία η Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι η κοινωνία μας αλλάζει λόγω ακριβώς αυτής της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας της κυβέρνησής μας. Συγκεκριμένα όταν λέτε εργάστηκαν για το άρθρο 8, για το κεφάλαιο συγγνώμη 8, θα σας πω δύο λόγια. Ο διάβολος δεν είναι στη λεπτομέρεια, αλλά στην εφαρμογή. Δεν αρκεί δηλαδή να υιοθετεί κανένα νομοσχέδια, αλλά να τα εφαρμόσει, να εφαρμόσει τους νόμους μετά και το λέω συνεχώς. Δεν αρκεί να ενσωμαθεί η κοινωτική νομοθεσία στην εθνική, αλλά να εφαρμοστεί κιόλα. Και στις 14 Δεκεμβρίου θα αξιολογήσουμε πόσο έχουν προχωρήσει, ιδίως και όσον αφορά την πρόοδο για το άρθρο 8. Τον λογισμό δηλαδή. Κύριε Κώστα, αναφερθήκατε στην ε, διαδικασία επανένασης της ε, Κύπρου. Εγώ ομολογώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθώ με τα θέματα που ε, ήταν στο τομέα των ομοιοτήτων μου. Δεν ήταν ο ρόλος μου να αναλάβω την εργασία των Ηνωμένων Εθνών που έχουν τη δουλειά αυτή εδώ και πολύ καιρό. Εγώ αναγκάστηκα να κοιτάξω στους έξι μήνες αυτός που είχαμε την Προεδρία πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ορμή του, τρένου της διεύνασης. Βέβαια, οι σχέσεις με την Τουρκία είναι σημαντικές για να υπάρξει μια ατμόσφαιρα, ε, σωστή ατμόσφαιρα για τις διαπραγματεύσεις. Πήγα βέβαια εγώ στη Λευκοσία, μίλησα με τον πρόεδρο Χριστοφιά. Εξετάστε να δω πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το δυναμισμό του προγράμματος και τις ενδεχόμενες λύσεις. Κατά βάση όμως, για να καταλάβω μόνο πώς θα μπορούσε η διαδικασία αυτή διεύρυνσης που ήταν η δική μου αρμοδιότητα να συνεχίσει να κινείται. Δεν πρέπει λοιπόν να αναμειγνύουμε τα πάντα και είναι σαφώς ότι όταν εξετάσουμε τη δική μου αρμοδιότητα εγώ εξέτασα ποια είναι τα κεφάλαια που μπορούν να ανοίξουν στη διαδικασία διεύρυνσης για την Τουρκία λαμβάνοντα πάντα βέβαια υπόψη ότι τα κεφάλαια που δεν είναι μπλοκαρισμένα πολιτικά παραμένουν, ε, γίνονται σιγά σιγά πολύ λίγα. Ακόμα δηλαδή και αν η Βελγική Προεδρία μπορέσει να αρχίσει ένα νέο διαπραγματευτικό κεφάλαιο που θα ήταν καλό, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα παραμένουν, θα γίνουν πολύ λίγα και χρειάζεται μια ειδική ορμή και ένα από τα στοιχεία για την καλύτερη ατμόσφαιρα είναι μια λύση βέβαια για την νήσο ή όπως είπατε πριν σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Και γι' αυτό συζητάω τα θέματα αυτά, πάντα βέβαια εν ώψη της προώθησης ανοίγματος κεφαλαίων. Δεν ήμουν δηλαδή υπερβοτικά φιλόδοξος και προσπάθησα να παρουσιάσω αυτόν σαν να είμαι κι άλλος εκπρόσωπος του ΟΗΕ ο καθένα έχει τη δουλειά του. Βέβαια είμαστε στην επαφή με εκείνου που έχουν αυτή την ευθύνη. Βέβαια, ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό η συμφωνία αυτή που είχε σαν στόχο να σταματήσει η βία. Και συμφωνώ με την αξιολόγηση της ε, Κομισιόν ότι η κυβέρνηση θα κάνει να κάνει περισσότερο για την εφαρμογή του και με ρωτήσετε ποιε είναι οι κύριε μου ανησυχίε. Εγώ ενδιαφέρομαι κυρίω στη διαδικασία αποκέντρωση και στην εξασφάλιση περισσότερη ε, διαφάνεια στι οικονομικέ δυνατότητε τη τοπική αυτοδιοίκησης και η καλύτερη συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Ε, καθορίσαμε λοιπόν κάποια στοιχεία που μας ανησυχούν. Για το ερώτημα Βεσνίας Ερζογοβίνης θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί ειλικρινά όταν συζητάμε για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 14 Δεκεμβρίου, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αποστείλουμε θετικά μηνύματα, να τονίσουμε ότι ο ευρωπαϊκός ρόλος αυτού του τμήματος του κόσμου είναι πραγματικά ευρωπαϊκός, αλλά ότι ακόμα πολλά μπορούν να γίνουν και προφανώς στις 14 Δεκεμβρίου δεν θα έχουμε σαφή πρόοδο. Το ίδιο ισχύει και για το κοσυφοπαίδιο. Γι' αυτό εισαγωγικά συζήτησα κάποιες από τις χώρες αυτές. Και τονίστηκε αυτό και όταν συναντηθήκαμε οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, υποθέσεων στο Σαράγεβο υπό Ισπανική Προεδρία το ακόμα. Για να πούμε ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν ένα ευρωπαϊκό στόχο αλλά δεν μπορεί να αντικαταστεί αυτό με το σκεπτικό ότι δώστε μας το χρονοδιάγραμμα να δούμε πότε θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να σε ενθαρρύνουμε στις προσπάθειές τους. Το θέμα της αναγνώρισης. Εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο που να αλλάζει ουσιαστικά την κατάσταση σήμερα. Ξέρετε ότι 22 χώρε έχουν αναγνωρίσει το 25, 5 δεν έχουν. Είναι βέβαια αληθέ ότι η επιτυχία και απαντώ εδώ και στον κύριο Σαραφράγκα που ρώτησε κατά πόσο πραγματικά η Λισαβόνα μα δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε με μία φωνή. Ναι, ναι. Από τσούμα, ναι. Στο ΝΟΙΕ, παραδείγματος το ψήφισμα για τη Σερβία, μιλήσαμε με μία φωνή και είχαμε μία ομοιόμορφη άποψη τα 27 κράτη-μέλη Ακόμα και να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πέντε από τις χώρες δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπέδιο και οι 20 το αναγνωρίζουν. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και δεν βλέπω να έχω αλλάξει άποψη σήμερα. Ούτε αυτές οι χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπέδιο έχουν αλλάξει ε, άποψη. Κροατία πόσα κεφάλαια. Και εδώ πρέπει να καταλάβετε το ρόλο μου ε, όταν είναι ένας τίμιος διαμεσολαβητής κάποιος ε, σημαίνει ότι καταβάλει τι καλύτερε δυνατές προσπάθειες για να πετύχει συνένεση. Είναι σωστό όμω να πούμε ότι θα εξετάσουμε προσεκτικά τουλάχιστον τρία κεφάλαια Ελπίζω να επιτύχουμε πρόοδο. Το δεύτερο ερώτημα πάλι για την Κροατία είναι κατά πόσον πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη της Ουγγρικής Προεδρίας θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την Κροατία. Αυτό που δεν πάρει σε μένα να γίνει δεν θα το επιβάλλω στο διαδοχό μου. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι στην Κροατία είναι επίσης ρεαλιστές. Αυτό που ακούω συχνά είναι ότι ορισμένα από τα πιο ενθουσιώδη ε, κράτη-μέλη επιμένουν για μια ε, ημερομηνία πολύ πιο νωρίς από εκείνη που λένε οι λογικοί άνθρωποι στην Κροατία. Γιατί κοιτάξτε, λέμε κεφάλαιο ανταγωνισμού, εύκολο να το πούμε. Αλλά περί τίνος πρόκειται, πρόκειται να κλείσουν ε, εργοστάσια, να σταματήσουν επιδοτήσεις του κράτους, χάνονται δηλαδή θέσεις απασχόλησης. Αυτά δεν είναι εύκολο λοιπόν να πραγματοποιηθούν και ε, συγχαίρω την κροατική κυβέρνηση για μια ανακοίνωση προς τον πληθυσμό πολύ ρεαλιστική όπου δεν προτείνεται κάποιες προθεσμίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το ρόδιμα να υποβληθεί καταρχήν στους κροάτες, τους ίδιους, γιατί ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει για να φτάσουν στο τέλος. Zeg me wat het probleem is. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik. <laughs> Diplomats want to protect me against myself, but there's no problem. να με προφυλάσει από αυτόν, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι πρόκειτο να μιλήσω, ε, να πω κάτι λάθος ε, ε, όταν θα μιλήσω για την τέος γεωκοσοφική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Κάτι άλλο είχα σημειώσει, αλλά ξέρετε, γελάτε ακούω. Α, ωραία αυτό. Well, um... Νομίζω ότι όλοι εσείς που λέτε ότι υπάρχει κάποια ανυπομονησία για πρώτα στο θέμα του ονόματος είναι αληθές νομίζω. Συμφωνούμε πολύ πάνω σε αυτό. ερωτήθηκε κατά πόσο ασκούμε πίεση. Ναι, ασκούμε πίεση, αλλά ισότιμα. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει κάποια συμμετρία, γιατί μια συμφωνία είναι μια ε, οδός διπλής κατεύθυνσης. Για το ταγκό δύο χρειάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συμφωνία για το θέμα των της ονομασίας και είναι σημαντικό για μας και για μένα να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και αν επιληθεί το θέμα της ονομασίας, πολλά θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να ενσωματωθεί το κοινωτικό κεκτημένο. Και κανένας δεν αποτρέπει μια χώρα να προσεγγίσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με το να προσαρμόσει την ομοθεσία της προς την Ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που λέω συχνά. Λένε πολύ ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που καταβάλλονται Τι γίνεται, μα κοιτάξτε, είναι ένα δώρο που κάνετε στους ε, πολίτες σας. Είναι θυσία να έχουν οι πολίτες σας κάποια ασφάλεια για τα τρόφιμα ή για, την, ε, για το κράτος δικαίου κλπ. Θυσία είναι αυτό ή δώρο. Νομίζω ότι να προσεγγιστεί το κοινοτικό κεκτημένο είναι κάτι που είναι πρόοδος για τη χώρα αυτή. Συμφωνώ με όλους εκείνους που μίλησαν για βοήθεια, ενίσχυση ε, προς τις χώρες αυτές στην οδό προς την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου. Αυτό γίνεται, δεν μπορώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες ίσως, διότι ο Επίτροπος Φίλε είναι εκείνος που οργανώνει αυτή την βοήθεια. Προς το τέλος υπήρχε μια καλή ερώτηση. Πώς θα μπορέσουν δηλαδή να ε, συνενωθούν οι προσπάθειες των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαδικασία αυτή διεύρυνσης. Κάποιος με ρώτησε, αυτή είναι η τελευταία φορά που η Προεδρία θα συζητάει το θέμα αυτό της διεύρυνσης. Όχι. Αυτό δεν είναι θέμα που θα ανατεθεί ποτέ στην ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεν είναι θέμα διπλωματίας, είναι κάτι το διακυβερνητικό. Και οι ε, εξαμηνές ε, προεδρίες θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να υπάρχει συνένεση μετά των κράτων μελών πώς θα μπορεί μια υποψήφια χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τώρα κατά πόσον μείναμε σε στενή επαφή με την ε, Κομισιόν, λέω ναι. Κατά πόσον έχουμε στενή επαφή με όλους τους παίκτες, αν θέλετε, με όλε τι πηγέ ε, επίδρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση είναι ναι. Αλλά θα παραμείνει το θέμα ε, ευθύνη της εξαμηνίας πρόεδρες. Η κυρία Κορνέλισεν αναφέρθηκε σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα όσον αφορά το κληροδότημα, είπατε, και τα μηνύματα στο 3 και πώς υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και ότι είναι δύσκολο τα κράτη-μέλη να μεταβιβάσουν αυτό το μήνυμα. Νομίζω και τώρα μιλάω εγώ σε εθνικός ε, πολιτικός ένα από, τα, με, από τις μεγάλες τραγωδίες είναι ότι οι εθνικοί πολιτικοί συνήθισαν να υπάρχει μια εύκολη διέξοδος. Όταν θέλει κανένας να μεταβάσει ένα κακό μήνυμα προς τους πολίτες, λέει φταίει η Ευρώπη. Αν θέλει να πει κάτι καλό, μπαίνει μπροστά στα φώτα της ράμπας και λέει αυτό πέτυχα, εκείνο πέτυχα ο τρόπος με τον οποίο η εθνική πολιτική μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικότατος για να πειθεί η κοινή γνώμη για αυτά που κάνουμε. Και βέβαια να τονιστούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η διεύρυνση είναι κάτι που πρέπει να ζητήσουμε να κάνουν οι εθνικοί μας πολιτικοί. Και η ιδέα σας για τον Δήμο που διευρύνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς να θέλω να πω ότι αύριο θα είναι πραγματικότητα αυτό. Για το κοσμοπέδιο. Εισαγωγικά νομίζω είπα ξεκάθαρα ότι εργαζόμαστε σε, πάνω σε μια προοπτική για να υπάρχει ένας διάλογος απελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίου και με το κοσυφοπαίδιο και η συμφωνία να υπάρχει μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οξυβοπηδίου. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένε ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηνύματα ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρό υπόψη την μοίρα των πολιτών του Κωσυφοπηδίου και ότι θέλουμε να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση που έχετε ήδη προτείνει. Το τελευταίο ερώτημα. Εγώ δεν θα σας ενημερώσω για τις προσπάθειές μου για να προσε... προσεγγίσουμε την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκερας. Αναφερθήκατε στη σκέψη ότι αυτή δεν θα είναι διαδικασία σταδιακή, αλλά θα πρέπει να είναι πραγματική. Δηλαδή, ή, εγώ διαφωνώ με την άδεια σας, διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές στην πολιτική πρέπει να γίνουν πραγματικά βήματα για να δημιουργηθεί μια νέα εμπιστοσύνη και να αλλάξει η διεύθυνση της ε, ε, συζήτησης οφείλεται πολλές φορές σε μια σταδιακή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να απάντησα σε όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ. Η συνάντηση νομίζω ήταν χρήσιμη, ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η φήμη σας για την ε, ειλικρίνειά σας αλλά και για το ευσύνοπτο των απαντήσεων σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνάντηση που είχαμε και ελπίζω να παραμείνουμε σε επαφή και να κρατήσουμε ε, τις επαφές αυτές με το Συμβούλιο και όχι μόνο με την είπα το εκπρόσωπο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto... Έχουμε λίγα λεφτά, πρωτοπορία στο ωράριο, προβλέπεται η ψηφοφορία στις 4.30 και χθε δεν ήταν δυνατόν να γίνει η συζήτηση για τα 4 και 5, έκθεση Κασίν δηλαδή, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κασίν για να ανακτήσουμε τον χρόνο που χάσαμε χθες. Έχετε το λόγο κύριε Κασίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης της ηγητές για την προσπάθεια που έκαναν. Μαζί τους καταλήξαμε σε 18 συμβιβαστικές, οι οποίες εντάσσουν, συμπεριλαμβάνουν θα έλεγα ένα μεγάλο κομμάτι των τροπολογιών. Η Κροατία προχωρά στις διαπραγματεύσεις. Το Μαυροβούνιο θα ανακηρυχθεί υποψήφια χώρα στο τέλος του μήνα. Γενικά έχουμε να κάνουμε με πολύ θετικές εξελίξεις για το σύνολο της περιοχής που δημιουργούν μια όθηση την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει και η Σερβία. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή, ό,τι φαίνεται, θα είναι η πιο θετική από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία και θα καταλήξει η διαδικασία αυτή στο να γίνει η Σερβία πλήρες μέλος της Ένωσης. Οι ευθύνε έχουν μεταφερθεί τώρα στον Αντιπρόεδρο Σβέτκοβιτς και θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του διαλόγου με την Πρίστινα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα του δικαστικού σώματος, της δικαστικής εξουσίας. Οι Σέρβοι λαμβάνουν υπόψη τα θέματα αυτά πάρα πολύ σοβαρά και ελπίζω να υπάρξει σημαντική πρόοδος στο μέλλον σχετικά με την εποκύρωση της ταφωνίας σταθεροποίηση με την Σερβία, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους τη σημασία της συμφωνίας αυτής για το σύνολο της περιοχής. Δίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες ένταξης ένα θα έλεγα ουδέτερο φόρουμ για συζητήσεις οι οποίες έχουν προσφέρει πολλά και θα προσφέρουν πολλά στη σταθεροποίηση της περιοχής. επικυρώθηκε από το, το Σερβικό Κοινοβούλιο χάρη και στις τροπολογίες των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης που δημιούργησαν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Αλλά λόγω της ανεπαρκούς συνεργασίας με το Διεθνές Δικαστήριο δεν ξεκίνησε η διαδικασία επικοινωνίας παρά μόνο τον Ιούνιο. Θα πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιπε 16 χώρες να επικυρώσουν τη συμφωνία με τη Σερβία το ταχύτερο δυνατόν. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διαδικασία των υποψηφίων και δυνητικά υποψηφίων χωρών. Μέσω της επικύρωσης της συμφωνίας με τη Σερβία ενθαρρύνουμε τη Σερβία να κάνει τα απαιτούμενα βήματα τα οποία δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν λόγω της επικύρωσης. Μετά και από τις προτάσεις του ε, Μπράμετς και στα πλαίσια της όθησης για το διάλογο στην Πρίστινα ελπίζω η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης να, να υπογραφεί σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Κατσίν. Έχουμε χρόνο για τρεις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Η κυρία Κοπά, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Κασίν, για μια θετική έκθεση για τη Σερβία, η οποία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Θα ήθελα επίση να το συγχαρώ και για τι συμβιβαστικές τροπολογίε. Η ομάδα μου πιστεύει ότι πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Σερβία για την πρόοδο που επετελέστη και γιατί ε, υπογραμμίζει τα προβλήματα τα οποία παραμένουν προς λύση. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει σύλληψη των καταζητουμένων και στα πλαίσια της έκθεσης ε, Μπράμετς. Η έκθεση αυτή τώρα για το κοσυφοπέδιο, η έκθεση δεν είναι για το κοσυφοπέδιο βέβαια, και το θέμα του κοσφοπεδίου δημιουργεί προβλήματα στα μέλη της Επιτροπής μας, μας διαιρεί θα έλεγα. η ομάδα μας επιμένει στις δύο συμβιβαστικές τοπολογίες 3 και 4 με τις οποίες συμφωνούμε και δεν θα υποστηρίξουμε άλλες τοπολογίες για τη Σερβία και θα ζητήσουμε και από τις άλλες πολιτικές ομάδες να κάνουν το ίδιο τέλος. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και θεωρούμε ότι έχει σημασία να στείλουμε ένα ξεκάθαρο ενιαίο μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας. Κυρία σε ένα λεπτό. Και εγώ θεωρώ πολύ θετική την προσπάθεια που έκανε ο κύριος Κασίν μέσω των συμβιβαστικών τροπολογιών. Υπάρχει το θέμα της συνεργασίας με το Διεθνές Δικαστήριο, όχι μόνο γιατί είμαι Ολλανδή, αλλά είμαι υπεύθυνη για την Βοσνία στην πολιτική μου ομάδα Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια σαφέστατη θέση. Ο Βλάντιτς και ο Χάρτιτς θα πρέπει να συλληφθούν πλέον. γιατί αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους θύματα του πολέμου και ε, δεν ε, θέλουν να αντιμετωπίσουν το παρελθόν με αντικειμενικό τρόπο. Ξέρετε ότι ετάφησαν εκ νέου 770 νεκροί του θύματα του πολέμου. Η Σερβία πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει τα πράγματα. Η έκθεση Μπράμετς τον προηγούμενο Ιούλιο δεν ήταν ιδιαίτερα θετική για τη Σερβία. Ελπίζουμε η νέα να είναι καλύτερη, αν και δεν υπάρχουν λόγοι για να μας οδηγήσουν σε αυτό. Υπάρχουν δύο έτη ακόμα περαιτέρω λειτουργίας του Διεθνούς Δικαστηρίου και η πλήρη συνεργασία με αυτό είναι βασικό κριτήριο για τη Σερβία. Συζητάμε τα θέματα αυτά και στη Συμβιβαστική 5 και οι περισσότερες ομάδες συμφωνούν να βγάλουμε τις λέξεις στα αγγλικά «the most». Μόνο η σύλληψη των δύο καταζητουμένων μπορεί να θεωρηθεί σαν πλήρης μορφή συνεργασίας. θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τις λέξεις the most και ε, ζητώ να μην ε, ε, και να δούμε με ποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει μπορούμε να αναδιατυπώσουμε την ιδέα αυτή. Καλώς. Κύριε Σόπφλιν και μαζί σας τελειώνει η συζήτηση. Ένα λεπτό. Πράγματι είναι πολύ καλή η έκθεση, νομίζω ότι οι συμβιβαστικέ τροπολογίες είναι καλές, δουλέψαμε σκληρά για αυτές. Να συγχαρώ τον κύριο Κασίν και συμφωνώ με όλα τα άλλα όσα ακούστηκαν. Καλώς, μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να ετοιμάσετε τις κάρτες σας. Ξεκινάμε με την πρόταση ψηφίσματος ε, για τη Σερβία και με τη Συμφωνία Συνεργασίας και Σταθεροποίησης. Παράγραφος 1, τροπολογία 19, υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 21, <clears throat> προφορική, ποιοι είναι υπέρ, κατά. 22 22 eh, προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 37. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. 41. Πρόκειται για ψηφοφορία κατά διέρεση. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα, τροπολογία της σοσιαλιστικής ομάδας, πρώτο τμήμα της τροπολογίας 41, ξεκινάει η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. 48 ψηφίζουν, μάλλον 47 ψηφίζουν, 24 υπέρ και 23 κατά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν την κάρτα και θέλουν να ψηφίσουν. Λοιπόν, 24 υπέρ, 23 κατά. Καλά, επαναλαμβάνω, ποιοι είναι υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, πρόεδρε, δεν έχω την κάρτα μαζί μου. Είμαι κατά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, ας, ποιοι είναι υπέρ πρώτα, παρακαλώ, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της 41. Εννοώ υπέρ αυτοί που δεν έχουν κάρτα όμως, όχι αυτοί που ψήφισαν ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ποιοι δεν έχουν κάρτα και θέλουν να ψηφίσουν, ποιοι είναι υπέρ. Τρεις, τέσσερις. Κοιτάξτε, καλά, δεν υπάρχει σύγχυση, θα πρέπει να ψηφίσουμε εκ νέου. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 41. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. 51 ψηφίσαντες. Για μια στιγμή. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να προσθέσουμε αυτούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, γιατί δεν έχουν την κάρτα τους. Μπορούν να σηκώσουν τα χέρια τους. Κύριε Τάνο, τι θέλετε. Διαδικαστικό. Δεν θέλω να υποπτευθώ κανέναν, αλλά δεν ξέρουμε αν οι μηχανές τους δουλεύουν ή όχι και δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε παρακαλώ την, μέσω της ανατάσεως των χειρών την ψηφοφορία. Γιατί κάποιοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν δύο φορές, λέει ο κύριος Στάνοκ. Πράγματι κάποιοι από τους συναδέλφους θα μπορούσαν να ψηφίσουν δύο φορές, είναι αλήθεια κύριε Τάνοκ. Εφόσον υπάρχει μία πιθανή συνωμοσία, ε όχι εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά νομίζω ότι μετά από την παρατήρησή σας δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σηκώσετε ψηλά το χέρι σας για να σας μετρήσουμε έναν προς ένα. Θα χάσουμε λίγο χρόνο για την τροπολογία 41. Ποιοι είσαστε του πρώτου τμήματος της 41 υπέρ. Και κρατήστε ψηλά τα χέρια σας γιατί πρέπει να σας καταμετρήσουμε σωστά.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 Λοιπόν, λοιπόν 27-27 δεν περνάει, καταπίπτει η τροπολογία. Δεύτερο τμήμα τώρα. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ του δευτέρου τμήματος. Όχι, δεν θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Περνάμε λοιπόν στην προφορική 1. Δεν ψηφίζεται η δεύτερη τροπολογία. Λοιπόν, προφορική παριθμένα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. δεκτή. Τροπολογία 51 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα της 51 υπέρ. Μας διακόπτουμε κυρία Λούνατσεκ. Πάντα στη 41. Τι έγινε με τη 41 λέει η κυρία Λούνετσεκ. Τι έγινε με τη 41. Λοιπόν, η 41 λέει ο πρόεδρος είχε διαιρεθεί σε πρώτο τμήμα, ε, ψήφισαν 27 υπέρ και 27 κατά και δεν έγινε δεκτό και το δεύτερο τμήμα δεν ψηφίζεται. Ψηφίζουμε τώρα το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 51. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ δεκτή. Το δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτό. 52 υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Σοσιαλιστική ομάδα ζητά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 52. Ξεκινάμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 24 κατά δεκτή, 53 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, συμβιβαστική 4 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, τροπολογία 55 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 5. Σε ξεχωριστά τμήματα, σύμφωνα με το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί, πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής 5, ποιοι είναι υπέρ, όλο το κείμενο εκτός από το λέξεις the most. Κυρία Κοπά, εμείς έχουμε αποσύρει το αίτημα ξεχωριστής ψηφοφορίας. Α, οι πράσινοι όμως επιμένουν. Καλώς. Βρισκόμαστε στη συμβιβαστική 5, το πρώτο τμήμα, όλο το κείμενο εκτέσα από τις λέξεις the most. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής 5, το πρώτο τμήμα κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα είναι υπέρ Κατά. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι είναι δεκτό και το δεύτερο τμήμα, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Για μια στιγμή, δεν σας έδωσα το λόγο κυρία Κορνέλισεν, δεν σας έδωσα το λόγο. Ζητήσατε το λόγο, δεν σας είδα, αλλά παρακαλώ ε, μη δημιουργείτε περαιτέρω σύγχυση το δεύτερο τμήμα. Δεν κατάλαβα πώς ψηφίσατε. Σας ζητώ λοιπόν να ψηφίσετε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Ο κύριος Τάνοκ. Κοιτάξτε, στον κατάλογο ψηφοφορίας, τουλάχιστον στη δική μου, στο δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας, θέλετε να μας πείτε πώς πρέπει να ψηφίσουμε, να κρατήσουμε το δεμόστο, το συν ή πλήνα. αυτός ο οποίος έχει καταθέσει την προφορική τροπολογία ή η γραμματεία μπορεί να μας εξηγήσει πώς ακριβώς θα ήθελα να ψηφίσουμε. Κοιτάξτε, η γραμματεία θα μας διαβάσει την τροπολογία. Λάβαμε το αίτημα από τους πράσινους να ψηφίσουμε το σύνολο της συμβιβαστικής 5 με την εξαίρεση των δύο λέξεων «the most». Λοιπόν, ψηφίσαμε το πρώτο τμήμα, το σύνολο του κειμένου, χωρίς τις λέξεις «the most» πριν από τη φράση «πιστικές αποδείξεις συνεργασίας» κτλ. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα αφορά μόνο τις δύο λέξεις, τα αγγλικά «the most». Για να επανέλθουν, αν θέλετε, οι δύο αυτές λέξεις στο κείμενο. Αν θέλετε το σύνολο της 5 πρέπει να υπερψηφίσετε και το δεύτερο τμήμα συνεπώς. Καλώς λοιπόν το δεύτερο τμήμα, συμβιβαστική 5 ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτή. 71. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 72 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 74 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές δεκτό 77 υπέρ Σοσιαλιστική ομάδα 76. Ψηφίζουμε το 76 ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. 32 κατά 22 υπέρ. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 89, 89 σε δύο τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές δεκτό το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβιβαστική 10 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 11 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 12 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 101 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. 102. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ 107 δεύτερο τμήμα κατά αποχές. Βέβαια, το αποτέλεσμα ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 107. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 17 κατά, 37 υπέρ, εγκρίνεται. 108. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 13 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 ποιος είναι υπέρ κατά Ε, Όχι, δεν ψηφίζουμε το 124. Πάμε κατευθείαν στη βαστική τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχισε, άρχεται η ψηφοφορία για την 135. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 33 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 138. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν βλέπω καλά τη διαφορά. Ψηφίζουμε με ηλεκτρονικό τρόπο την τροπολογία 143. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 31 ψήφισαν υπέρ και 24 κατά εγκρίνεται. 144. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 ποιος είναι υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158. Προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Α. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Ή μάλλον όχι, καταπίπτει. 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa la Τέλος ψηφοφορίας ψήφισαν 40 υπέρ και 17 κατά. Γιατί δεν σηκώνατε τα χέρια σας υπέρ, άρα εγκρίνεται. 14, ποιος είναι υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17, ποιος είναι υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. 15, μάλλον όχι, καταπίπτει. 16, ποιος είναι υπέρ. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Με βάση τις ενδείξεις των συντονιστών, κανονικά θα πρέπει να έχει εγκριθεί, αλλά δεν σηκώστε τα χέρια. Συμβαστική τροπολογία 18 ή καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση. Καλά. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 18. Δεύτερο τμήμα, τροπολογία 18, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 υπέρ 15 κατά, αλλά μόνο οι συντονιστές σηκώνουν τα χέρια. Εν πάση περιπτώσει, συμβαστική τροπολογία 18, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τρία, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε στην 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. «51 υπέρ 3 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έγινε δεκτή η πρότασή του με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα έχουμε μία, μία, μία μονή ψηφοφορία για την σύσταση την σχετική πάντα με τον κύριο Κατσίν. Ποιοι είναι υπέρ. αν πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία και εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Λοιπόν, 51 ε, υπέρ, 0 κατά, 2 αποχές, μεγαλύτερη πλειοψηφία, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 5-6 ε, λεπτά διακοπή πριν από τη συνάντηση και κλεισμένων των θυρών με τον πρέσβη Έγκερερ. Σε 6 λεπτά ε, ξεκινάμε πάλι.